κάθε φορά πριν τις ψηφοφορίες. Εγώ θέλω να τηρήσουμε το πρόγραμμά μας και να ακούσουμε και τα καταληκτικά σχόλια στο τέλος της συζήτησης για τα κατεπήγοντα. Λοιπόν, θα παρακαλούσα τώρα τον κύριο Τάνοκ να πάρει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ζάμπη είναι από τις λίγες χώρες στην Αυρική όπου έχουμε πάνω από δύο ειρηνικές παραδόσεις παραλαβές της εξουσίας από το 1991 με πολυκομματικές εκλογές. Πέρυσι έγιναν εκλογές και ο πρόεδρος Λούγκου κέρδισε με μικρή διαφορά τον Χακαΐντε Χιτσιλέμα. Και ε, τώρα υπάρχουν ανησυχίες. Ε, το συνταγματικό ε, δικαστήριο ε, ε, απεφάνθη κατά του Χιτσιλέμα και πρόσφατα τον έχουν συλλάβει και τον έχουν κατηγορήσει για προδοσία. Δικτατορία που δεν λέει το όνομά της χαρακτηρίζει και ο επίσκοπος ε, την κατάσταση. Ο πρόεδρος προσπαθεί να εκαθιδρύσει την εξουσία του, όπως έχουμε δει ε, και ο πρώην, τον πρώην πρόεδρος Σιλούμπα να ε, προχωρήσει το 2001 σε μια τρίτη θητεία αντισυνταγματική. Τώρα θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πέσουν οι τόνοι και η Ζάμπια να υποστηριχθεί και στο ευρωπαϊκό, συγγνωμη, δημοκρατικό τη ε, σύνταγμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κοράου για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατηγορείται για εσχάτη προδοσία. Υποτίθεται ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα γιατί η αυτοκινητοπομπή του προσπέρασε την αντίστοιχη του Προέδρου Τσιλούμπου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιμετωπιστεί η αντιπολίτευση στην ε, ε, Ζάμπια. Δυστυχώς υπάρχουν συλλήψεις, βασανισμοί και νομίζω ότι η δύναμη μιας κυβέρνησης είναι το να δέχεται και να επιτρέπει την κριτική εις βάρος της. Νομίζω ότι ο κύριος Τσιλέμα και όσοι συνελήφθησαν μαζί του θα πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και θα πρέπει να ξεκινήσει μια έρευνα έτσι ώστε να δούμε αν πράγματι έχει υπάρξει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπό το φως των τελευταίων συμφωνιών συνεργασίας θα πρέπει να δούμε τι οικονομική βοήθεια δίδουμε εμείς ε, στην κυβέρνηση Λούγκου έτσι ώστε να μην υπάρχει παραβίαση των κοινοτικών κανόνων. Post. Η Ζάμπια για πολλά χρόνια είναι μια από τις περισσότερων υποσχόμενες χώρες. Υπήρξαν δύο ειρηνικές μεταβάσεις πολιτικές, αλλαγές πολιτικές ε, στην εξουσία, κάτι το οποίο είναι σπάνιο στην Αφρική. Τώρα όμως ε, τα πράγματα φαίνεται να έχουν αλλάξει και ε, η κυβέρνηση ε, κατηγορείται για αυταρχικές συμπεριφορές. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης έχει σύλληφθεί με ψευδεπίγραφες κατηγορίες. Η σύλληψη του κυρίου Χατζηλίμα όμως είναι η κορφή του παγόβουνου. Η κοινωνία των πολιτών υποφέρει ε, έχει πολιτικοποιηθεί πλήρως η δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε να ε, βλέπουμε ότι η Ζάμπια οδεύει προς την δημοκρατία. Ο πρόεδρος Λούγκου θα πρέπει να γνωρίζει ότι τον παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε. Επόμενο μιλήτρια, κυρία Σένρα Ροντρίγες. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λαμβάνοντα υπόψη τη σημερινή κατάσταση στη χώρα, θέλουμε να κάνουμε έκκληση στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση για να αρχίσουν ειρηνικό και επικοδομητικό διάλογο, προκειμένου να ξεπεραστούν οι πολιτικέ εντάσει που υπάρχουν σήμερα και για να επικεντρωθούν στη λύση των μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που πλήττουν τον λαό του. Η φτώχεια στην Ήπεθρο το 2015 ήταν 76,6% Τρει φορέ παραπάνω από ό,τι στι πόλει. Και δεν υπήρξε μείωση από το 2010 μέχρι το 2015. Το πρόβλημα της διατροφής είναι υπεύθυνο για 54% των θανάτων των παιδιών. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Το UBVH, το AIDS δηλαδή, είναι ενδημικό στη χώρα. Γι' αυτό και ζητάμε από τις αρχές να προωθήσουν τα δικαιώματα των πολιτών και τα πολιτικά τους δικαιώματα και να φροντίσουν να υπάρξει δίκαιη αντιμετώπιση στον Χακάιν Τεχιτσιλάμε βάσει των διαφόρων αφρικανικών και διεθνών ε, συμφωνιών. Έτσι θα σταματήσουν αυτή την ε, διακριτική μεταχείριση σε βάρος πολλού. Διακόπτη ο Πρόεδρος, πρέπει να τηρούμε το χρόνο μας γιατί δεν έχουμε χρόνο. Βέντα, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ και τις άλλες πολιτικές ομάδες για την καρποφόρα συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας, συντάσσοντας το ψήφισμα αυτό. Το 2016 στην προεκλογική εκστρατεία υπήρξαν ήδη πολιτικές εντάσεις ανάμεσα στο κόμμα, ε, στην εξουσία και στην αντιπολίτευση. Η Ζάμπια βέβαια έχει πετύχει πολλά μεταβάσεις πολιτικές οι οποίες έλαβαν χώρα σε καθεστώς ειρήνης. Τώρα όμως ο Χιτσλέμα, ο κύριος ηγέτης της αντιπολίτευσης, δεν αναγνωρίζει την νίκη του Προέδρου Λουγκού εξού και συνελήφθη και κατηγορείται για προδοσία. Κάτι που σημαίνει ότι τον περιμένει θανατική ποινή. Αυτό είναι ο κίνδυνο. Παρόλο που τα τελευταία 20 χρόνια δεν υπήρξαν εκτελέσεις στη Ζάμπια, θεωρητικά η θανατική ποινή παραμένει. Ισχύει. Και πιθανόν να ε, υλοποιηθεί, δεδομένου ότι μιλάμε για προδοσία. Έχουμε βέβαια πληροφορίες ότι οι λόγοι για τους οποίους διώκεται το χιτλέμα είναι πολιτικός. Ε, είναι πολιτική μάλλον και όχι τίποτα άλλο. Γι' αυτό και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει πολιτικό διάλογος με τις δύο πλευρές με την δικιά μας στήριξη, τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Πρέπει να υπάρξει δίκαια δίκη. Πρόεδρος. Πήγα να σας διακόψω, συγγνώμη όμως, γιατί τηρήσατε το χρόνο σας. Καλώς. Τώρα, μισή λεπτό, κύριος Μαρίνιο. Ευχαριστώ ο αγώνας μας υπέρ των θεμελιδών δικαιωμάτων, στην περίπτωση της Ζάμπια για παράδειγμα, απαιτεί δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να ενισχυθούν οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Και πρέπει επίσης να διευρυνθεί και το πεδίο δράσης του ακόμα και σε χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη της Ρώμης κανένας υπεύθυνο δεν πρέπει να παραμένει ατιμόρυτος. Αυτό είναι το καλύτερο που έχουμε να προσφέρουμε στα θύματα τέτοιων παραβιάσεων. Γιατί είναι αποτρεπτικό στοιχείο. Και το κύριο, κυριότερο αποτρεπτικό στοιχείο που διαθέτουμε. Τα άλλα μέτρα που θα έπρεπε να πάρουμε είναι πολιτικής και οικονομικής φύσης. Και απαιτούν να δώσουμε πραγματικό αγώνα κατά τις φτώχειας. Γιατί όπου υπάρχει φτώχεια πάντα θα υπάρχει για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η φτώχεια από μόνη της αποτελεί παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Οι εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων, ο κύριο Πρέντα, για ένα λεπτό εξ ονόματο του ΕΛΚ. Oh, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο ήταν εκείνη που ζήτησε να γίνει αυτή η συζήτηση για τη Ζάμπια. Υπάρχουν εντάσεις από την εποχή ε, των προεδρικών εκλογών, από πέρσι το καλοκαίρι. Και οξύνθηκε η πολιτική κρίση μετά την ε, σύλληψη του ηγέτη της αντιπολίτευσης Χιτσιλέμα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δεινή ο άνθρωπος κινδυνεύει να του επιβληθεί η θανατική ποινή για μια παράβαση του ΚΟΚ. Υποτίθεται ότι παρεμπόδισε την αυτοκινητοπομπή των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενοχλεί ο κύριος Ιτσιλέμα γιατί τόλμησε να αμφισβητήσει τις προεδρικές εκλογές, το αποτέλεσμά τους δηλαδή. Αλλά βασικά αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να συζητάει με την αντιπολίτευση, όχι να τη διώκει. Σοσιαλιστέ και δημοκράτε, η κυρία Κιέγγε, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα την δυνατότητα να ηγούμε της Επιτροπής Εκλογικής Παρατήρησης στη Τζάμπια. Θέλω να ευχαριστήσω την Φορντερίκα Μογκερίνη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Δεν αρνούμε ότι συναντήσαμε δυσκολίες στην εκλογική διαδικασία και περιορισμού στην ελευθερία έκφρασης, ε, μικρή συμμετοχή των γυναικών, κακή λειτουργία του συνταγματικού δικαστηρίου. Όμως το αποτέλεσμα είναι σωστό. Ε, ο τέος πρόεδρος υπερίσχυσε του υποψηφίου της αντιπολίτευσης εμείς λοιπόν αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης ε, στη Ζάμπια και γι' αυτό η απελευθέρωση του κυρίου Τσίτσιλέμα θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία επίδειξη σεβασμού της δημοκρατίας και της πολιτικής εναλλαγής και θα είναι ένα παράδειγμα και για τις υπόλοιπες χώρες της Αφρικανικής Υπήρου. Ο κύριος Σαφοζέρ Συνάδελφοι, προφανώς και πρέπει να ανησυχούμε για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζάμπια. Απ' την άλλη τίθεται ορισμένα ερωτηματικά. Όταν κάποιος λειτουργεί κατά της ασφαλείας της χώρας και το θέμα της προδοσίας το έχουμε δει και στις δικές μας χώρες στο παρελθόν, να συνδέεται ε, με θέματα ασφαλείας και στη Γαλλία και στις Ηνωμένε Πολιτείες χρησιμοποιήθηκαν οι κατηγορίες αυτές για να αποσταθεροποιηθούν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Παρεμβαίνουμε στο όνομα των αξιών μας, μα οι αξίες μας θα έλεγα αμφισβητούνται, γιατί με δύο μέτρα και σταθμά κατηγορούμε τους άλλους και τι κάνουμε εμείς. Εμείς τι κάνουμε, η Κίνα τι κάνει, η Ινδία τι κάνει. Αυτές οι χώρες δεν παρεμβαίνουν σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερα για τη Ζάμπια όπως και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν εσωτερικές αντιφάσεις δύσκολες. Πρέπει να αντιμετωπίσει την αστικοποίηση, τον εξυγχρονισμό της, τον εκδημοκρατισμό της, τον τόσο δύσκολο, σε ένα κλίμα διεθνούς ανταγωνισμού που απαγορεύει την δημιουργία ενός σωστού οικονομικού ιστού υπό την επίβλεψη του ΔΝΤ. Συνεπώς λοιπόν στην ουσία άγεται και φέρεται η Ζάμπια θα πρέπει να αφήσουμε λοιπόν την διάσκεψη των τοπικών επισκόπων και τον Οργανισμό Αφρικανικής Ενότητας να βρουν λύσεις επί τη βάση της αρχής της επικουρικότητας και μόνον αυτής. Ευχαριστώ συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε τώρα με τη διαδικασία του Catch the Σας ευχαριστώ να σεβαστείτε αυστηρά το ένα λεπτό. Ο πρώτος ο μιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια Ο κύριος Χιτζηλέμα, ο επικεφαλής ε, της αντιπολίτευσης, κατηγορήθηκε για προδοσία και συνελήφθη. Αν προσθέσουμε σε αυτό και τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης στη χώρα, ε, αυτά είναι τα στοιχεία που βλέπουμε από την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας. Η αποχρησιμοποιούν οι αστυνομικοί, ε, ο κίνδυνος φυλάκισης με ισόβια ή και θανατική ποινή είναι πράγματα που απειλούν το κράτος δικαίου και τις διεθνείς υποχρεώσεις στη Ζάμπια. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταδικάσει κάθε προσπάθεια εκφοβισμού των μελών της αντιπολίτευσης και να αρχίσει διάλογος ανάμεσα στο ε, κόμμα της ε, κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης ώστε να επιστρέψει η δημοκρατία στη Ζάμπια. Ευχαριστούμε, Γραπίνη. Τώρα για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Πίτροπε, η κατάσταση στη Ζάμπια είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθούμε στενά. Πρέπει να συνεισφέρουμε και εμείς έναν ειρηνικό και επικοδομητικό διάλογο και χαιρετίζω τη δέσμευση των τοπικών εταίρων. Εγώ πήγα στη χώρα και είδα τη φτώχεια που επικρατεί και το φόβο για την επόμενη μέρα. Πρόκειται για ανθρώπου. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε διεθνή επίπεδο υπέρ τη δημοκρατία και τη απάλληψη τη φτώχεια. Εξάλλου θανατική ποινή εξακολουθεί να ισχύει στη χώρα αυτή, κάτι που είναι απαράδεκτο. Και υπάρχει και περιορισμός στην ελευθερία έκφραση που μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσει. Γι' αυτό ακριβώ θα ήταν πάρα πολύ καλό το ψήφισμα αυτό να τεθεί σε εφαρμογή. Ο κύριο Μαριά, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ζάμπια είναι μια φτωχή αφρικανική χώρα η οποία πραγματικά αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα και λόγω της εξάπλωσης του aids. οι συγκρούσεις που διαμορφώνονται μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης οφείλονται στην αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών τον αύγουστο του 2016, όταν και ο πρόεδρος λούγκου κέρδισε με πολύ μικρή διαφορά έτσι η αμφισβήτηση εκ μέρους του χιτζιλέμα δηλαδή του αρχηγού της αντιπολίτευσης έχει οδηγήσει σε συγκρούσεις έχει συλληφθεί ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και κινδυνεύει ακόμη και η ζωή του. είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. νομίζω ότι και η ευρωπαϊκή ένωση η κομισιόν πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό για να αποκατασταθεί η ηρεμία στην περιοχή να μπορέσουν οι δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις να βρουν μια λύση διότι το κυρίαρχο πρόβλημα στη ζάμπια είναι η φτώχεια. αυτό πρέπει να δουν και με βάση αυτό το γνώμονα να λύσουν τις διαφορές τους. ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριος Καστάλντο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν μπορεί κάποιος να κατηγορηθεί για σκάτη προδοσία επειδή εμπόδισε μια προεδρική το πομπή Μπορεί να σας φαίνεται αυτό αδύνατο, αλλά στη Ζάμπια συμβαίνει. Ε, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης διώκεται γι' αυτό το λόγο. Και μάλιστα ε, συνελήφθη με κάποιους συνεργάτες του μαζί και κατηγορείται για εσχάτη προδοσία. Επίσης, ε, και άλλοι κρατούνται και κατηγορούνται για εσχάτη προδοσία Μπορεί να έχουν γίνει ε, κάποιες ατασταλίες στις εκλογές. Δεν είχαμε ουσιαστικά όμως την δυνατότητα να ελέγξουμε την τελική καταμέτρηση πριν αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο το εκλογικό. Εμείς θέλουμε η Ζάμπεα να απελευθερώσει τον Χιτσιλέμα και τους συνεργάτες του, να σεβαστεί τη Συμφωνία του Κοτονού και να σταματήσει αυτή τη φάρσα λόγω της οποίας κινδυνεύει με θάνατο ο κύριος Χιτσιλέμα. Να θυμίσω ότι 488 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με πολύ σωστό τρόπο σε σχέση με την περιοχή αυτή. Ο κύριος Πόλτσακ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ε, ήθελα να ευχαριστήσω τους συντάκτες ε, αυτού του ψηφίσματος γιατί ε, πραγματικά επέστησαν την προσοχή μας σε αυτή τη χώρα. Καμία πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί. Υποτίθεται ότι θα προχωρούσαν. Αν δούμε τι έγιναν στις προεδρικές εκλογές, λένε και οι παρατηρητές των εκλογών ότι δεν ήταν όλα πρόσκοπτα και κανονικά. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης ε, έχει συλληφθεί, ε, κρατείται και αυτό είναι απαράδεκτο. Τώρα θα κληθεί ε, να δοκιμαστεί η Ζάμπια για να δείξει ότι υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και σέβεται η χώρα τη διάκριση των εξουσιών. Εμείς θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τη δίκη αυτή, να δούμε αν είναι δίκαιη και αν η Ζάμπια ε, ανταποκρίνεται ε, στην πραγματικότητα και στην πρόοδο που έπρεπε να έχει γίνει. Η Επίτροπος παρακαλώ για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, έχω τη χαρά να μιλώ εξ τη κυρία Μογκερίνη. Σα ευχαριστώ για αυτή την επίκαιρη συζήτηση για τι εξελίξει στη Ζάμπια αξίζουν πραγματικά την προσοχή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά πάρα πολύ τη συνεργασία της και την εταιρική σχέση με τη Ζάμπια και είναι και περήφανη για τη συνεισφορά στην ανάπτυξη της χώρας. Είμαστε στεναρά προσιλωμένοι ε, στην εταιρική μας συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει επίσης τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και υποστηρίζει ε, τους φιλόδοξους οικονομικούς στόχους και ε, το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Θυμάστε ότι είχαμε στείλει και παρατηρητές στις εκλογές την ηγεσία της κυρία Σισελ Κέγκε που μίλησε προηγουμένως εκτιμούμε πάρα πολύ και ευγνωμονούμε την κυρία Κέγκε για την εργασία της αυτής. Έχουν κάνει συστάσεις ιδιαίτερα σχετικά με τις ανησυχίες για την ελευθερία της έκφρασης και ε, του συνέρχεστε. Η Ζάμπια παραδοσιακά ήταν μια χώρα ειρηνική και δημοκρατική σε μια γειτονιά που πολύ ε, συχνά ε, σπάραζόταν από ε, πολιτική αστάθεια και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό μας ανησυχεί ε, πολύ που αμφισβητείται η δημοκρατική πορεία της χώρας. Ιδιαίτερα από τον Αύγουστο του 2016 και τις προεδρικές εκλογές που ήταν πάρα πολύ αφιλεγόμενες και πόλωσαν πάρα πολύ τα πράγματα στη χώρα. Η σύλληψη του ΧΑΚΑΙΝΤΕ Χισιλέμα στις 11 Απριλίου ε, όξινε ακόμα περισσότερο τις πολιτικές εντάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ωστόσο ανταποκρίθηκε αμέσως, ζήτησε από όλες τις πλευρές να σταματήσουν οποιαδήποτε πράξη ή ε, ρητορική που ε, οξύνει την κατάσταση. Σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουμε να στέλνουμε αυτό το ισχυρό μήνυμα και προς την κυβέρνηση και προς την αντιπολίτευση έτσι ώστε να διαδραματίσουν επικοδομητικό ρόλο και να αρχίσουν ένα διάλογο για να επανέλθει η εμπιστοσύνη και η υποστήριξη ε, της ε, πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς σε σχέση με τη δίωξη του κυρίου Χισιλέμα και τη δίκη, καλούμε την κυβέρνηση της Ζάμπιας να εξασφαλίσει ε, διαφάνεια στη δίκη, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη με τις δικονομικές εγγυησει σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Οι θεσμοί της χώρας θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Είναι πολύ σημαντικό για να διατηρηθεί η δημοκρατία και η πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους τη Ζάμπια μέσω όλων των διάβλων πολιτικών και διπλωματικών σε όλα τα επίπεδα και ε, απευθυνόμαστε στο αίσθημα ευθύνης όλων έτσι ώστε να ε, σεβαστούν την ισχυρή δημοκρατική παράδοση στη Ζάμπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση για τη Ζάμπη.